μέλλον, αλλά να μην βαδίζουμε προς το μαύρο μέλλον, το ζωφερό μέλλον, να βαδίσουμε προς ένα ε, ανοιχτόχρωμο μέλλον με ελπίδες. Σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Επόμενο σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη ε, είναι η προφορική ερώτηση εξ ονόμου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς την Επιτροπή και αφορά στο έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Ίδωρ. Το λόγο έχει ο συντάκτης ε, κύριος Ρίχαρντ Ζέιμπα για πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Προετοιμάζουμε ένα ψήφισμα για το φόρουμ το οποίο θα λάβει αυτήν την εβδομάδα στη Μασαλία. Δυστυχώς ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν ε, να συμμετάσχουν και δεν συμμετείχαν γιατί ήδη ξεκίνησε, γιατί τρέχει η Ολομέλεια. Θέλω όμως να σε επισημάνω ότι πρόκειται για το έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ και να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ήδη ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του 2010. Ένα ψήφισμα το οποίο επιλαμβάνεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαίωμα στο το νερό ε, στις ε, εγκαταστάσεις υγιεινής. Αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά μας. Όμως θα μου επιτρέψει να σε κάποιους αριθμούς ε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στη γη έχουμε 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αλμυρό νερό. Και αυτό το 2,5 μόνο αυτού είναι το ε, γλυκό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βρίσκονται στα υπόγεια ύδατα. Κατόπιν τούτου για την ανθρώπινη κατανάλωση έχουμε πάλι μόνο το 1% αυτού, δηλαδή 200.000 ε, κυβικά χιλιόμετρα και το 60% αυτή τη στιγμή ήδη χρησιμοποιείται. Αν δούμε λοιπόν ότι η κατανάλωση του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο επίπεδο ε, διπλασιάζεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να ε, διερωτηθούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα το νερό. Με βάση τα στοιχεία των μέτρων περίπου το 70% χρησιμοποιείται για την υδροδότηση στη γεωργία, το 22% στη βιομηχανία και 8% στα νοικοκυριά. Επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έντονη αστιφιλία ε, κυρίως στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες και οι προβλέψεις ε, λένε ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο μέχρι το 2050 θα έχουμε αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 50%. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία θα δούμε ότι το 2050 κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε 9,3 δις ανθρώπους στη γη, 70% ε, περισσότερα τρόφιμα σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλες θα είναι οι ανάγκες νερού νερού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και ε, θετικά μηνύματα ως ε, ε, πρώτη το στόχο της χιλιετίας αναφέρουμε την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό το πετύχαμε και αναφέρεται στην τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Ε, το 2015 θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Δυστυχώς ε, στις εγκαταστάσεις υγιεινής δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε με σαφήνεια ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να πετύχουμε τους στόχους μας, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του νερού, τότε θα πρέπει να έχουμε σαφή πολιτική και εξέλιξη. Γιατί ε, ας μην ξεχνάμε ότι ε, και στην Ινδία και στην Κίνα υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς ε, και στη Βόρεια Αφρική, στη Μαύρη Αφρική κυρίως, που δεν υπάρχουν πολλά θετικά μηνύματα. Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα θετικό είναι ε, το νήμα που διατρέχει αυτό το έκτο ε, φόρουμ που είναι Time for Solutions, έτσι λέγεται. Έχουμε λοιπόν θεσπίσει πολλά ψηφίσματα, τώρα έχει φτάσει η χρονική στιγμή τα ψηφίσματα αυτά να υλοποιηθούν. Το Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού ε, θέλει, πρόκειται να επεξεργαστεί 12 προτεραιότητες με τρεις στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, η διασφάλιση ευημερίας των ανθρώπων. Δεύτερον, ο πλανήτης να παραμείνει μπλε και τρίτον ε, να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Τι καλούμεθα λοιπόν να πράξουμε για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Εμείς εκφράζουμε τις απόψεις μας στο ψήφισμα και πιστεύω ότι είναι σημαντικό καταρχήν να βελτιωθούν τα στοιχεία. Ε, υπάρχει τεράστια έλλειψη όσον αφορά τα ουσιαστικά στοιχεία για το νερό. Ε, ποιοι είναι οι καταναλωτές, ποια είναι η ρήπανση και πάρα πολλά άλλα. Να βελτιωθεί λοιπόν η συλλογή των δεδομένων για να μπορούμε να χαράξουμε σωστή πολιτική. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τους ποταμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό να σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει και σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι καθοριστική σημασία οι χώρες που έχουν κοινά σύνορα να συνεργάζονται. Ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται συγκρούσεις ε, λόγω του νερού. Εδώ υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Η συνεργασία είναι ευκαιρία για να διαφυλαχθεί η ειρήνη. Καθοριστική σημασία είναι επίσης ε, να ληφθούν στο μέλλον σωστέ αποφάσεις για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, λαμβάνοντα υπόψη το νερό. Αυτό αφορά τη βιομηχανία, αφορά τη γεωργία και τη βιομηχανική παραγωγή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τελειώνω κύριε Πρόεδρε το ότι το νερό έχει και ένα έντονα τοπικό χαρακτήρα. Σε ορισμένε περιοχέ. υπάρχει έντονη λειψιδρία, σε άλλε πάλι όχι. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ο κύριος Ποτότσνικ, ο συναδελφός μου, δεν μπορεί να βρεθεί, να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Γι' αυτό τον αντικαθιστώ με μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ συμμετείχα στο έκτο φόρουμ υδάτων μαζί με τους συναδέλφους Πι και Γεωργίεβα. Θα ήθελα να σας πω ότι η Γαλλία που μας φιλοξένησε. Στη Γαλλία συντάξαμε την κοινή μας ανακοίνωση και ξέρετε ότι φτάσαμε σε μια συνεκτική πολιτική υδάτων. Από το 2000 με την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων μιλάμε για ένα πολύ καλό στάτους μέχρι το 2015 των υδάτων με την καλή διαχείριση του πλαισίου. Έτσι όλοι οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ε, εξουσία πέρα από τα εθνικά καθαρά όρια. Παρά τις προσπάθειές μας όμως οι στόχοι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί διότι υπάρχουν θέματα διαχείρισης που σχετίζονται με την ποιότητα και ποσότητα υδάτων θα πρέπει να δούμε τις περιβαλλοντικές αλλαγές, τις κλιματικές αλλαγές και να δούμε κατά πόσο λαμβάνουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές στην πολιτική μας περί υδάτων. Στο φόρουμ παρουσιάσαμε μια κοινή πλατφόρμα εμείς που αποτελεί μια συγκεκριμένη λύση ως προς την, τους υδάτινους πόρους για να αντιμετωπίσουμε και τις πλημμύρες. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας για να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων της χιλιετίας. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα, στους υδάτινους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Αυτό το προσχέδιο, το blueprint, ορίζει δράση σε 7 τομείς. Οι οικονομικά κίνητρα για να δούμε πώς θα προβούμε στην τιμολόγηση των υδάτων, αποδοτικότητα για να βρούμε μία εργαλειοθήκη και μέσα για τη στοχοθέτηση τον, το, για τη στοχοθέτηση ως προς υδάτινους πόρους, επίσης εταιρική σχέση δημόσιου ιδιωτικού τομέα, επίσης το προσχέδιο θα ορίσει την διακυβέρνηση και το ε, διοικητικό πλαίσιο για να φτάσουμε σε μια σωστή ε, τεχνογνωσία. Καλύτερα στατιστικά στοιχεία για να δούμε πώς ε, προωθούνται και πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους πόρους καθώς και έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θα ε, ενισχύσουμε τα μέτρα μας στον τομέα της υγείας και υγιεινής ως προς το πόσιμο νερό η νέα μας πολιτική στη διαχείριση των υδάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αφορά συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης με βάση τις ε, δικές μας πρωτοβουλίες. Η Υπουργική Δήλωση συμπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για αλλαγές τονίζοντας τους βασικούς στόχους περί υδάτων. Λίγει ο κύκλο των ομιλητών εξ των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει εξ ονόματος κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο Χριστιανοδημοκρατών η κυρία Σοφή Οκονή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα της πρόσβασης στο νερό και στο καθαρό νερό είναι βασικό για όλους μας. Είναι ο λόγος για τον οποίο Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ένωσα τις δυνάμεις, δυνάμεις μου με τον συνάδελφο Ρίτσαρντ Μπέρ για να ετοιμάσουμε ένα ψήφισμα. Πράγματι, μέσω του νερού μιλάμε για τις συνθήκες υγείας και επιβίωσης χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων. Έρχομαι από το Μπουρκίνα Φάσο που δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό. Έζησα μέσα στα τέλματα, ζήσα τις δυσκολίες του λαού, την ανασαχή, ανησυχία τους και την αρρώστια των παιδιών. Χαίρομαι λοιπόν που ο πρώτος στόχος της χιλιατηρίδας του ΟΗΕ υλοποιήθηκε πριν από το 2015, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει νερό διαιρέθηκε δια δύο από το, 2000, ε, από το 1990 μέχρι το 2010. Θαυμάσιο νέο, αλλά έκκληση για δράση επίσης. Η επιτυχία ποτέ δεν τελειώνει. Χαίρομαι λοιπόν για αυτό το ψήφισμα και ειδικότερα αναφέρομαι σε τρεις βασικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα, όπως σας το είπα, Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους της χιλιοδηγίδα του ΟΓΕ, ειδικότερα όσον αφορά το καθαρό νερό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης τη διαχείριση του νερού αναδεξαμενή γεωγραφική και η επεξεργασία πρέπει να γίνεται ανάντι και όχι κατάντι. Ακόμη πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση όλων των λαών στο νερό. Σας μίλησα για την Πουρκίνα Φάσο. Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Σέρμπου Ντατσιάνα Οκτάβια. Για, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η πρόταση ψηφίσματος διαβιβάζει ένα σαφές μήνυμα στο Διεθνές Φόρουμ Ιδάτων. Θα πρέπει να μην θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα εμπόρευμα που ε, παράγει ε, ε, κέρδος αποκλειστικά. Πρόκειται για βασικό δικαίωμα του ανθρώπου και γι' αυτό θα ήθελα να διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα στα, στη Μασαλία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιηθεί το είδος στη γεωργία. Το 70% όπως ξέρουμε χρησιμοποιείται σε γεωργικές δραστηριότητες και σε ορισμένες χώρες αυξάνεται στο 80 έως 90%. Άρα η πρόσβαση στο νερό ε, είναι ύψιστη της σημασίας και γι' αυτό θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες της διατροφικής αλυσίδας. Για να φτάσουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις νέες τεχνικές, να υποστηρίξουμε τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να άρουμε και τα προσκόμματα από τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70% του ύδατος ε, κινείται, μάλλον μεταφέρεται στη γεωργία και το 30% το χρησιμοποιούμε για τη διατροφή. Γι' αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο Ίδωρο για λόγους διατροφικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει επίσης η βιοποικιλότητα και οι κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την πλήρη αντιμετώπιση αυτού του θέματος και ελπίζω να διαβιβαστεί αυτό το μήνυμα στη Μασαλία καθώς και στη διάσκεψη του Ρίο. Η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ο κύριος Γκέρμπεν Γιάν Γκερμπράντι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εφόσον πρόκειται για το νερό και για το πόσο σημαντικό είναι το νερό σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, πολλές φορές ε, παρατίθενται απόψεις ε, του Διευθυντή των ΗΕ που είπε ότι η πόλεμη, η μελλοντική πόλεμη θα είναι για το νερό. Δυστυχώς λοιπόν αυτή είναι μια πρόβλεψη που έγινε παλαιότερα και επαληθεύτηκε ή επαληθεύεται. Πολύ συχνά ε, ξεχνάμε πολλά πράγματα. Ο ίδιος άνθρωπος είπε ότι ε, εάν δεν υπάρξει ε, καλύτερη διαχείριση αυτού του βασικού αγωθού θα έχουμε ε, ολέτρια αποτελέσματα. Το νερό πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Και στη Μασαλία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα συζητηθεί και τον Ιούνιο ε, στη συνάντηση Ρίο Αυτή την εβδομάδα δημοσιεύτηκε η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ε, και αυτός είναι ανησυχητικός. Δεν είναι όμως ε, η τοπαθής. Ε, περιέχει βέβαια ε, κριτική, αναφέρει ότι υπάρχει υπερβολική χρήση του νερού στην Κίνα, στη Μέση Ανατολή, στην Καλιφόρνια. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ε, πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό, όπως και με το ρόλο που παίζει η γεωργία στην εξάντληση των υδάτινων πόρων. Υπάρχουν και άλλα θέματα σημαντικά. Εχθές η Δανική Προεδρία συνομολόγησε μια συμφωνία με την Κίνα για τη μεγαλύτερη εξαγωγή τεχνολογίας στην Κίνα. Τα επόμενα 10 χρόνια η Κίνα θα επενδύσει 500.000 εκατομμύρια στη διαχείριση των υδάτων γιατί το νερό είναι και οικονομικός παράγων. Ε, στο Ρίο λοιπόν πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση νερού στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Η κυρία Μισελ Ριβαζή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα καλό, ένα θετικό πρώτα απ' όλα ε, σε σχέση με το ψήφισμα για το νερό. Ε, Καταδεικνύει τις καλές προθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη διαχείριση του νερού. Ε, γίνεται λοιπόν αυτό το Διεθνές Φόρουμ. Ξέρετε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Προέδρου, του Λουίντε Φουσόν, που είναι και πρόεδρος των ε, ε, λουτρών της Μασαλίας. Δηλαδή είναι περισσότερο φόρουμ εμπορικό και όχι διεθνούς συμφέροντος. Δηλαδή ε, υπάρχει μια τάση των συλλογικών οργανών να θέλουν να αποκτήσουν πάλι τη διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων. Λοιπόν, το φόρουμ αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να κατευθύνουν τη σωστή διαχείριση του νερού. Και αυτό είναι μια τάση ιδιωτικοποίησης και για την Ευρώπη και για τις χώρες ΑΚΕ. Τώρα, ε, νερό και υγεία. Ε, ξέρουμε ότι το μη πόσιμο νερό όταν ε, το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οδηγεί σε ασθένειες και πραγματικά πρέπει να επενδύσουμε στην επεξεργασία των αποβλήτων ε, και των βιομηχανικών λιμάτων που αποβάλλονται χωρίς επεξεργασία στη φύση. 70% είναι αυτό του συνόλου νερό και ενέργεια. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε βεβαίω το νερό και ξέρετε ότι το θέμα του σχιστόλιθου και των αερίων των σχετικών μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο υπόστρωμα και μπορεί να οδηγήσει σε μαζική ρήπανση. Τσακωνόμαστε λοιπόν για την ποιότητα του νερού, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Miroslav Για Ευχαριστώ. Θεωρείται πολύ συχνά ότι επικρίνω την περιβαλλοντική μας πολιτική. Αλλά στην περίπτωση των υδάτων θα ήθελα να πω ότι θα υποστηρίξω τους προλαλήσαντες. Τα ύδατα αποτελούν ένα διεθνές πρόβλημα και η κακοδιαχείρισή τους θα οδηγούσε σε ολέθριες συνέπειες. Γι' αυτό υποστηρίζω την διάσκεψη η οποία έχει ξεκινήσει και το προσχέδιο ψηφίσματος με ε, ορισμένες μικροαλλαγές. Αναφέρεται ότι πρόκειται για έναν ε, βασικό πόρο της ανθρωπότητας και δεν θα πρέπει να είναι πηγή κερδούς. Ε, αν υποστήριξουμε αυτή την πρόταση, νομίζω ότι θα ε, υπάρξουν κίνδυνοι στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό υποστηρίζω την ε, τροπολογία του κυρίου Ζέμπερ και άλλων να μιλήσουμε για παράνομο κέρδος. Και εάν περάσει αυτή η τροπολογία θα υποστηρίξω ολόκληρη την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η Στάλφος ε, Ματίας ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι στην Πορτογαλία με ευρωπαϊκά κονδύλια και μη έχουμε φτάσει σε ένα 98% ε, και 90% αντιστοίχως κάλυψης στην παροχή υδάτων και τον τομέα της υγιεινής. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα του τι προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα των υδάτων σε εμάς, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δηλαδή μη θεωρούμε το, τα ύδατα ένα εμπόρευμα. Είναι ένα, ε, ένας ο οποίος τίνει να εκλείψει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να κατασπαταλούμε τα, το νερό. Το, τα ύδατα είναι ένα βασικό δικαίωμα και δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε επικερδές εμπόριο. Δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα. <clears throat> Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πάσκα. Κύριε Επίτροπε, το νερό είναι πολύ σημαντικό για τον πλανήτη μας. Ε, το χρειαζόμαστε για τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία, την οικονομία. Η επάρκεια σε νερό ορίζει το που μπορεί κανείς να ζήσει και που μπορεί να καλλιεργήσει προϊόντα. Ε, έχουμε προφήτες ε, που είπαν για ότι το νερό έχουν μια μαγική δύναμη στη ζωή. Βέβαια, οι ποσότητες συντάτων είναι περιορισμένος. Η κατανάλωση αυξάνεται και επειδή δεν δημιουργούνται νέες πηγές υδάτων πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε αποτελεσματικότερα και να προστατεύουμε την ποιότητά του. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ε, υπάρχει και νομοθεσία για αυστηρή χρήση των υδάτων. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει σωστή χρήση στη βιομηχανία, κυρίως έτσι ώστε να μην σπαταλιέται ούτε μία σταγόνα νερό. Ευχαριστούμε. Ο Σνάλφος Στάτλερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, οι μέχρι τώρα ε, συνεδριάσεις ε, του Παγκόσμιου Φόρουμ του ε, Νερού καθορίστηκαν από τις προσπάθειες να υπάρξει σωστή διαχείριση των υδάτων και το στηρίζουμε. Είμαι ευγνώμων στην Ζέμπερ που στηρίζει και αναφέρει την οδηγία του 2000 όπου προβλέπεται η χρήση υδάτων τις εκβολές ε, ποταμών. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το ότι πρέπει να υπάρχει εξοικονόμηση δάτων και αυτό να επιβραβεύεται. Και απευθύνομαι στην κυρία Επίτροπο. Υπάρχουν πολλά κράτη που εδώ και 12 χρόνια στην εφαρμογή της ε, οδηγίας πλαίσιο δεν επιδεικνύουν πειθαρχία. Από το 2009 είχαν τα κράτη να εφαρμόσουν την οδηγία αλλά δεν συνέβη αυτό ε, και εδώ και τρία χρόνια και η δική μου χώρα παραβιάζουν ε, αυτές τις οδηγίες. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την ε, κυρία Επίτροπο αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στο φόρουμ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην οδηγία περί υδάτων. Ε, σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι ε, το ψήφισμα αυτό είναι σε γενικές γραμμές σωστό, σωστό το μήνυμα που εκπέμπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έκτο φόρουμ υδάτων και κατόπιν του εγώ θα υπερψηφίσω την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστούμε κύριε Στάτλα ε, και τώρα έχουμε ε, τους επόμενους αγορητές, καταρχήν τον κύριο Σόνικ. Πρόεδρε, νομίζω ότι πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται ότι 40% της ανθρωπότητας δεν έχει πρόσβαση στο νερό. Αυτά είναι τα στοιχεία και δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν νερό που δεν είναι πόσιμο, είναι ανθυγιεινό, και το νερό βεβαίω είναι απόλυτα απαραίτητο για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει συνεπώς να εξοικονομήσουμε το νερό. Έτσι θα καταπολεμήσουμε και τη φτώχεια. Επίσης, η πρόσβαση στο καθαρό νερό είναι βασικό, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Έχει αναγνωριστεί από την Παγκόσμια Διακήρυξη και από πολλά άλλα έγγραφα. Τέλειωσε ο καιρός όπου είχαμε εύκολη πρόσβαση στο νερό. Πρέπει συνεπώς να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που υφίστανται δημογραφικά πλέον. Έχουμε πληθυσμούς που ενισχύονται συνεχώς. Δεν πρέπει να το ξεκινάμε αυτό, πρέπει να συζητάμε το ζήτημα να αναγνωρίζουμε την κατάσταση και να ευαισθητοποιούμε με τη σειρά μας την κοινή γνώμη. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων σε αυτό, παγκόσμια, γιατί μόνο με μια τέτοια υποστήριξη θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε Σόνικ, ο κύριος Παρνιό για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή ε, Επίτροπο, σε σχέση με αυτό το ψήφισμα, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ασχοληθώ με δύο ζητήματα. Αφενός στη διαχείριση του νερού και αφετέρου έχω και μία ερώτηση για την Κομισιόν σε σχέση με ενέργειες για να ανταποκριθούν στο ενδιαφέρον μας μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Την πρόκληση δεν ξέρουμε. Το νερό είναι η μεγάλη υπόθεση του 20ου. Επειδή θα έχουμε απαντήσεις θα έχουμε και ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε τι είναι οι για τη διαχείριση, για την ασφάλεια των τροφίμων. Και σε σχέση με αυτό το φόρουμ, όπως το υπενθύμισε και ο συνάδελφος Ριβαζή, ε, δυστυχώς ενεπλάκησαν πολλά ενδιαφέροντα εμπορικά στη συζήτηση που γινόταν στη Μασαλία με στο πλαίσιο αυτού, αυτού του φόρουμ. Γιατί δεν υπάρχει τώρα συνοχή, συνέπεια μεταξύ διαχείρισης του νερού και ΚΑΠ. Τίποτα στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν καταδεικνύει ότι θα υπάρξει μία διαχείριση όπως την υπογράμμισε ο συνάδελφος Σαρμπού. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, συνάδελφο κύριος ε, Γκιούρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η σπουδαιότητα του θέματος και η σχετικότητά του με την ανάπτυξη θα έπρεπε να είχε, είχαμε συμμετάσχει περισσότερο στην προετοιμασία αυτής της συζήτησης. Βεβαίω το νερό είναι ένα σπάνιο είδος, είναι ε, βρώμικο, δεν είναι πόσιμο κτλ. κτλ. Ε, σε όλες τις εταιρικέ σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει το νερό να είναι ένα θέμα συζήτησης. Για κάθε ζήτημα, και αν, για οποιοδήποτε ζήτημα και αν πρόκειται, δεν είναι εμπόρευμα το νερό. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζονται ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην παραβιάζεται το νερό. Ο κατασκευαστής ο οποίος φτιάχνει τις κατάλληλες υποδομές ε, για το νερό και ο βιοτέχνης ο οποίος φροντίζει να μην υπάρχουν ροές τις οποίες δεν, δεν καλύπτει όλοι κατατείνουν προς την ίδια κατεύθυνση δηλαδή το γενικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Φερέρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Ιούλιο του 2010, μετά από μία μακρά μάχη, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ένα ψήφισμα και είπαν ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Γι' αυτό θα θέλαμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Δεν ήταν εύκολο να εγκριθεί αυτό το κείμενο και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα κράτη-μέλη έθεσαν βέτο και απέσχον στην τελική ψηφοφορία. Γι' αυτό θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πολύτιμο αγαθό. Όλοι έχουν ε, δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό. Δεν πρόκειται για, θέμα, ε, για ιδιωτικό θέμα, αλλά για ένα κοινό αγαθό. Ευχαριστούμε για μισή λεπτό, κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα διότι το ε, νερό δεν είναι μία ανανεώσιμη πηγή. Ε, μέρη ανανεώνεται μόνο, αλλά δεν ε, επανέρχεται στο ίδιο σημείο από όπου ε, ξέρευσε. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και τα ποτάμια ύδατα θα πρέπει να τύχουν σωστής διαχείρισης. Και το βλέπουμε και στην περίπτωση της Τουρκίας που δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένα ε, δεδομένα ως προς τον ε, ε, υδάτινο ορίζοντα. Δεν πρέπει λοιπόν να μην λάβουμε υπόψη την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Θα πρέπει να αλλάξουμε την θεώρησή μας ως προς την αντιμετώπιση της γεωργίας, γιατί δεν μπορούμε να καταβάλουμε άλλο αντίτιμο για την κατανάλωση ε, δηλαδή στον γεωρικό τομέα άλλο νερό χρειάζεται για το μαρούλι και άλλο για τον αραβόσιτο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εστέλα για ένα λεπτό. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ποσότητα και την ποιότητα του ύδατος και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των ε, κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μου στο τέλος του Φεβρουαρίου το 68% του εδάφους βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας και 32% σε, σε, σε κατάσταση απόλυτης ξηρασίας. Η κρίση των υδάτων ως προς την ποιότητα και την ποσότητα αφορά τη χρήση και την κατάχρηση των φυσικών πόρων. Πρόκειται και για θέμα διαχείρισης. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό σύστημα υδάτινης διαχείρισης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανεπάρκειες ως προς το 50% της διαχείρισης των υδάτων. Το νερό θα πρέπει να μην υπόκειται στο αλόγιστο κέρδος θα πρέπει να μην γίνεται και κατασπατάληση των υδάτων. Ευχαριστούμε κυρία Στρέλα. Η κυρία Βερζιά για 1,5 λεπτό. Για ένα λεπτό. Το έκτο φόρουμ υδάτων δεν αποτελεί μοναδική πλατφόρμα διαλόγου. Το θέμα είναι ότι όλοι ε, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα ύδατα. Πρόκειται για έναν πόρο ο οποίος είναι αναγκαίος για τη ζωή και όχι μόνο για τους ανθρώπους. Δεν ανήκει στον άνθρωπο. Είναι ένα κοινό, δημόσιο αγαθό. Μιλάμε για τη διαχείριση αυτών των υδάτων και η εταιρική σχέση, ιδιότητα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τις ευθύνες μας έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αλόγιστο κέρδος. Χαίρομαι διότι στη Γαλλία πολλές, πολλοί δήμοι και κοινότητες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του ύδατος, των υδάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διαδικασία ε, Catch the Eye. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Νικολεύκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι το 2050. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το είδωρ στις γεωργικές εκτάσεις, γιατί ήδη το 70% χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν την χρήση στη γεωργία με νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι θα πρέπει ίσως να γίνει μεγαλύτερη ε, χρήση γενετικός τροποποιημένων οργανισμών, διότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν σε είδωρ. Ευχαριστούμε πολύ και ακολουθεί η συνάδελφος κυρία Σμόλκοβα. Πρόεδρε, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές περιοχές του, χώρου, του κόσμου. Από την άλλη, εμείς ε, που έχουμε το νερό πολλές φορές ε, δεν το χρησιμοποιούμε ορθολογικά, το σπαταλάμε και αυτή λοιπόν η κακή διαχείριση του νερού οδηγεί στο ότι αλλάζει το κλίμα. Αν λοιπόν μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις εκπομπές ε, καυσαρίων και την βιομηχανική παραγωγή, τότε ε, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και καλύτερα τα υπόγεια ύδατα ε, και θα μπορέσουμε επίσης να επιτύχουμε και την παρακράτηση υδάτων στο έδαφος. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε λιγάκι και για τις υδάτινες οδούς ε, γιατί κάθε χρόνο δημιουργούνται πολλά προβλήματα ε, ζημιές ε, υλικές αλλά και ζημιές σε ανθρώπινες ζωές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν οφείλει να λάβει μέτρα έτσι ώστε το νερό να παγιδεύεται εκεί που βρίσκεται να φτάνει στις ρίζες των φυτών και να εμπλουτίζει τις πηγές. Ακολουθεί η συνάδελφος Μιράντα. Ευχαριστώ. Προέρχομαι από το Ντός όπου ο μεγάλος μας ποιητής μιλούσε για τα ποτάμια και τις πηγές. Δυστυχώς όμως ιδιωτικοποιήθηκε η διαχείριση υδάτων ε, και ο υδροφόρος ο ορίζοντας συρρυκνώθηκε και δυστυχώς και οι δατοφράκτες αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής διαχείρισης. Θα πρέπει να αλλάξουμε, να μιλήσουμε για βιωσιμότητα. Δεν πρόκειται για ένα ε, αγαθό ε, που οδηγεί σε κέρδος. Είναι μια, ε, ένας δημόσιος πόρος. Είναι ζωή στη ζωή θα πρέπει να προστατεύσουμε την ποιότητα των υδάτων, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του υδροφόρου ορίζοντα των ε, ποταμών, των θαλασσών και ούτω καθεξής. Sinclair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον διεθνή διάλογο στη Μασαλία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί που αποφασίζουν να προωθήσουν πραγματικά δυνατότητες για το νερό. Το νερό είναι κοινό αγαθό, απαραίτητο και βεβαίως είναι και ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί για υπερβολικό εμπορικό ε, κέρδος. Ο Λουί Φωσόν πράγματι έχει δημιουργήσει κάποιες συζητήσεις και πρέπει να, ε, τα κράτη να ε, ενισχύσουν την αποθοκευτική τους δυνατότητα. Η Ένωση των Γεωργών του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άμεση λύση και στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, όπως είπε και συνάδελφος, δεν αναφέρεται το ζήτημα του νερού Δηλαδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει με μία γλώσσα και ξεχνάει τα ζωτικά θέματα. Κυρία Γιόρνταν τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ζωή των ανθρώπων είναι άρρητα συνδεδεμένη με το νερό. Δεν μπορούμε να περάσουμε τη μέρα χωρίς το νερό. Όσον αφορά δε, την τροφοδοσία, δεν έχουμε ασχοληθεί πραγματικά με αυτό το ζήτημα. Επαρκώς τουλάχιστον. Στην Ευρώπη πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι βέβαια πολίτες δεν ε, ζουν ε, αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως τρίτες χώρες με πολύ φτωχούς ανθρώπους και ακόμη και προχωρημένες κοινωνίες λόγω της ενίσχυσης του πληθυσμού της αποψήλωσης και της μία ανάπτυξης σιγά σιγά θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα αν συνεχίσουμε να το παραμελούμε. Ε, στη Σλοβενία, τη χώρα μου, από την άποψη του νερού πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Όμως εμφανίστηκαν ε, περίοδοι ξηρασίας και αντιμετωπίζουμε προβλήματα και είναι σίγουρο ότι πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρότατα. Η συνάλφος Κλάς για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ε, Catch the Eye. Οι συγκρούσεις ε, για το νερό καθιστούν ε, σαφή τη σοβαρότητα της κατάστασης. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Παρ' όλα αυτά 900 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και 2,6 δις ε, άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινές εγκαταστάσεις. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι θεμελιώδης δικαίωμα και όλοι πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα. Η πολιτική μας πρέπει να βασίζεται στην αρχή του εφοδιασμού και της αρχή αρχής της υπετιότητας. Πρέπει να αποφύγουμε την διασπάθηση. Η μεταφορά τεχνολογίας για καινοτομία στον τομέα του νερού και της επεξεργασίας νερού πρέπει να προαχθεί. Πάνω από 90% των λιμάτων από τη βιομηχανία και τα ε, νοικοκυριά ε, διοχετεύονται ε, σε υδάτινους δρόμους. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν τεχνολογίες για να επεξεργαζόμαστε τα λίματα αυτά. Το καθαρά καθαρό νερό και οι υγιεινές εγκαταστάσεις είναι το κλειδί για το μέλλον και στη Μασαλία πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο κυρία Κλάς. Ε, η, κυρία, η Επίτροπος έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. First, Mrs. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα να διευκρινίσω το ότι η Επιτροπή ε, δεν ε, έχει αμφισβητεί το ότι ε, πρέπει να υπάρχει ένα νομικό καθεστώς. Αυτή λοιπόν η επιλογή εξαρτάται και από τα κρατημέλη. Ο κύριο Στάτλε αναφέρθηκε σε προβλήματα που έχουν σχέση με την οδηγία πλαίσιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρόσφατα συνήλθαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και είχαν μια ουσιαστική συζήτηση για το ότι είναι απαραίτητο στην Ευρώπη να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή. Όταν λοιπόν ε, θα αναφερθεί το αποτύπωμα στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή ε, νομίζω ότι θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η νομοθεσία στην Ευρώπη. Και τέλος ε, αναφέρθηκε ότι το νερό ε, θα είναι όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται στην κοινή οικιακή πολιτική έμεσα στον πυλώνα ΔΙΑ. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Πανιού πολύ σωστά λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει με τους αρμόδιους επιτρόπους και πρέπει να σας πω ότι το θέμα θα ε, επανέλθει στον κύριο Ποτότσνικ και στους άλλους επιτρόπους όπως πολύ σωστά το ζητήσατε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την ε, ε, κυρία Επίτροπο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση και κατατέθηκε πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος